Πρώτο σημείο, δήλωση της Επιτροπής για την ολοκλήρωση της ενίας ψηφιακής αγοράς. Παρακαλώ κύριε Μπαρνιέ. Πρόεδρε καλημέρα. Καλημέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πρώτο σημείο σημερινή διατάξης. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υποστήριξή τους σε μια πάρα πολύ σημαντική διαπραγμάτευση που ολοκληρώθηκε στο Μαρακέσε με ένα σχεδόν ομόφωνο ψήφισμα για την πρόσβαση ε, των εμποδιζόμενων ως προς την όραση ατόμων ε, στα βιβλία. Ήταν δυσχερέστατες οι διαπραγματεύσεις ε, και ολοκληρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα και εσείς ψηφίσατε, όπως είπα, σχεδόν ομόφωνα το ψήφισμα για αυτό το ζήτημα. Είχαν αναλάβει εξάλλου προσωπική δέσμευση εξ Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα να σας πω ότι σημειώνεται μεγάλη πρόοδος για την Ευρώπη των πολιτών, που είναι και ο στόχος μας. Δεν απέχουμε πολύ από την ενιαία ψηφιακή αγορά με ε, πελώριο δυναμικό. Η, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνει πρόοδο κατά 10% σε σχέση με τις ευρυζωνικές ε, συνδέσεις, θα, θα κερδίζαμε μια ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ, εάν το ηλεκτρονικό εμπόριο αντιστοιχούσε στο 15% του συνολικού εμπορίου, ε, αντί για το 5% που ισχύει τώρα, θα κερδίζαμε 1,7% ως προς την ανάπτυξη Ξέρουμε ότι 2,6 ε, ε, θέσεις απασχόλησης δημιουργούνται για μία που χάνεται χάρη στη ψηφιακή αγορά θα πρέπει λοιπόν να το επιδιώξουμε, όπως είπε ο Μάλκομ Χάρμπουρ και τα μέλη της Επιτροπής του που κατέχουν αυτό το ζήτημα, σε αυτό το επιχείρημα που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια, ε, δηλαδή τις πράξεις για την ενιαία ψηφιακή, για την ενιαία αγορά μάλλον. Εδώ και τρία χρόνια επεξεργαζόμαστε αυτό το νέο κανονιστικό αλλά δυναμικό πλαίσιο για να αναπτύξουμε την ενιαία ψηφιακή αγορά. Εγγράφεται δε η δράση μας ε, στην ε, συνέχεια προηγουμένων ε, οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών παραδείγματο χάρη και αναμένεται η μεταγραφή στην Εθνική Νομοθεσία για το τέλος του τρέχοντος. Αυτό ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών επιγραμμικά και άρα στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Τα τελευταία τρία χρόνια ε, ενεγράφησαν όλα αυτά σε μια συνολικότερη στρατηγική, δηλαδή τη συνολικότερη φιλοδοξία της στρατηγικής της συναδέλφου Ε, και έχουμε την πράξη μιας αγοράς ε, ένα και δύο θα επανέλθω σε αυτό και έχουμε και το στοχοθετημένο πρόγραμμά μας ε, για τις εμπορικές συναλλαγές και τις υπηρεσίες στην ενιαία ψηφιακή αγορά που μας απασχολεί στην Επιτροπή σε συνδυασμό και με την Ελικρός και με τον νέο συνάδελφο τον Κροάτη ο κ. Μπίμητσα. Έτσι προσεγγίσαμε το στόχο μας, ε, ο οποίος είναι η ψηφιακή αγορά που είναι και το βασικό μας ατού μεσούσης της κρίσης, ε, να λειτουργήσει πιο εύρυθμα και να ολοκληρώσουμε την ψηφιακή επανάσταση. Επισκόπηση υπεπραγμένων. Υπάρχουν τρία βασικά νομοθετήματα για τα οποία καταλήξαμε σε κοινή συμφωνία με το Συμβούλιο Εποργών. Υπάρχει ο κανονισμός ε, για τις ε, διαφορές ε, ως προς τους καταναλωτές που εγκρίθηκε τον Απρίλιο, τη οδηγία για τα ορφανά έργα και στη συνέχεια το Connect Europe Facility, νέο χρηματοδοτικό μέσο συνδέοντας την Ευρώπη. Στις 27 Ιουνίου καταλήξαμε συμβαστική λύση. Βεβαίως το κονδύλι υπολείπεται σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με τις αρχικές ε, προσδοκίες και φιλοδοξίες μας. Αυτά για τα πεμπραγμένα δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες. Συνέχεια ε, προϊούσε συζητήσεις ε, για συγκεκριμένες προτάσεις, δυναμικές επίσης, προτάσεις κανονισμού σε σχέση με τις πωλήσει και το κοινό δίκαιο για τις πωλήσει. Ο κύριος Λένε και, και ο κύριος Μπέρλιγκερ είναι αρμόδιοι. Στη συνέχεια ηλεκτρονικό εμπόριο και υπηρεσίες εμπιστοσύνης εισηγητή η συγγήτρια είναι η κυρία Ούσκο. Ε, πρόταση κανονισμού για την προστασία των δεδομένων. Ο κύριος Κέλλην, ο εισηγητής σας. Ε, σημαντικό διακύβευμα για την εμπιστοσύνη στη ψηφιακή αγορά. Η οδηγία για τον εξυγχρονισμό της συλλογική διαχείρισης της Μαρή Γκαλό για τις πολυεδαφικές υπηρεσίες και στη συνέχεια μείωση του κόστους για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών, πάλι εδώ η κυρία Χέρτζοκ, και κατόπιν ε, ηλεκτρονική τιμολόγηση. Βάσει των αναλύσεών μας, αξιότιμοι βουλευτές, ε, το γεγονός και μόνο θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε την ηλεκτρονική τιμολόγηση μας προσφέρει σε αυτή την ενιαία αγορά δύο, ε, επιπρόσθετα δύο δις μέχρι το τέλος του τρέχοντος ε, και με το τέλος της κοινοβουλευτικής ε, θητείας σας ε, θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει. Αυτό ελπίζουμε. Τώρα τα επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια. Ashley Fox. έκθεση πρωτοβουλία Γιώργαν Κρόιτσμαν για το ίδιο ζήτημα, στρατηγική για την πληροφορική, για το υπολογιστικό νέφος, το cloud computing. Η κυρία Αντελκαστή Γιοβέρα είναι η αρμόδια και κατόπιν ε, ένας ε, μεγάλος φάκελος ε, του οποίου επιλαμβάνει το κύριο Σφάμπ για την κυβερνοασφάλεια. Σε σχέση τώρα με την κατασκοπική δράση των ΗΠΑ, της οποίας έχει πέσει θύμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από την προστασία από πλευράς άμυνας, κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να αναζητήσουμε και μία απάντηση, κυρίως σε καιρό κρίσης. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κατοχυρώσει τη στρατηγική της ε, αυτονομία. Ε, και δύο είναι τα βασικά στοιχεία, ε, υπολογιστικό νέφος και κυβερνοασφάλεια. Υπάρχει όμως το Γαλιλαίο επίσης με τη δυνατότητα να προστατεύσουμε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών. Ιδού, όλα αυτά επιτάπητος. Είναι πολύ άριθμοι φάκελοι, πάρα πολύ σκληρό το έργο μας και ε, μας περιμένουν σημαντικές εξελίξεις, αυτά αναφέρετε και εσείς στο ψήφισμά σας, όπου ο Πάμπλο Αρία ε, Ετσεβάρια με την υποστήριξη του Μάλκομ Χάρμπορ κάνουν σοβαρέ προσπάθειε για να προωθήσουν το ηλεκτρονικό εμπόριο. Έχουμε πλήρη επίγνωση αυτή τη σκληρή πραγματικότητα και γι' αυτό θα επικεντρώσουμε τι προσπάθειέ μα σε τρει στρατηγικού άξονε και από αυτόν έχουμε καταθέσει και προτάσει. Το δυναμικό του ηλεκτρονικού εμπορίου πρώτα απ' όλα με μία ε, ε, δημόσια διαβούλευση ω ήθιστε. Έχουμε αναλάβει δράση για δύο βασικού τομεί που εντοπίσαμε στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Πρώτα απ' όλα θα προτείνουμε στι προσεχεί εβδομάδες φιλόδοξο εξυγχρονισμό των αγορών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών. Θα βασιστούμε στις συστάσεις ε, της έκθεσης κυρία Τερό. Ε, μέσα στο πακέτο αναθεώρηση τη οδηγία ε, για τις ηλεκτρονικές πληρωμές καθώ και μία πρόταση νομοθετικού περιεχομένου ρεαλιστική σε σχέση με τις ε, προϋποθέσεις ε, διασύνδεσης για να μπορέσουμε να τονώσουμε τον ανταγωνισμό, να διευκολύνουμε την πρόσβαση των καταναλωτών, αλλά και εφόσον μιλάμε για τους καταναλωτές, ε, να προσφέρουμε περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες ως προς τις πληρωμές, καθώς και να διασκεδάσουμε τις θεμίτες ανησυχίες και φόβους που υπάρχουν. Το φθινόπωρο στη συνέχεια θα προτείνουμε ένα αποτελεσματικότερο και ελκυστικότερο σύστημα για την ε, διακρατική μεταφορά και παράδοση προϊόντων που έχουν παραγγελθεί επιγραμμικά. Πάλι ο κ. Τσεβαρή είναι υπεύθυνο για να διευκολύνουμε και του καταναλωτέ αλλά και τι επιχειρήσει, κυρίω τι μικρόμεσε, που θέλουν να αναπτύξουν τι επιγραμμικέ διασυνοριακέ πωλήσει του και να δημιουργηθεί αυτό το φαινόμενο της διασύνδεσης, ε, ε, οι διασυνοριακές παραδόσεις αγαθών κοστίζουν ε, το τριπλάσιο ή πενταπλάσιο ποσό για αντίστοιχες αποστάσεις και 70% των επιγραμμικών παραγγελιών εγκαταλείπονται λόγω προβλημάτων παράδοσης. Θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση και κάνουμε μια ευρεία διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για αυτές τις διασυνοριακές παραδόσεις και κυρίως με τους ταχυδρομικούς φορείς οι οποίοι έχουν δηλώσει στην πρόθεσή του να σημειωθεί πρόοδο σε αυτό το τομέα. Δεύτερο βασικό άξονα, εξυγχρονισμό για τα δικαιώματα του δημιουργού και του σχετικού κανονιστικού πλαισίου. Δεν θα πρέπει λοιπόν να αντικαταστήσουμε ούτω ή άλλω την ε, ουσιαστική παραδοσιακή κατανάλωση. Ε, είναι άειλα πλέον τα προϊόντα και αυτό απειλεί ε, τον τομέα της δημιουργίας. Ε, έχουμε βασιστεί στο δίκαιο της εδαφικότητας μέχρι τούδε και αυτή τη στιγμή κινούμεθα μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον που δεν γνωρίζει σύνορα. Ε, τα δικαιώματα δημιουργού δεν πρέπει να αποτελέσουν φραγμό στην, εμπορική, στην ανάπτυξη του εμπορίου και να παρεμποδίσουν ναι, και την ανάπτυξη αλλά και την καινοτομία. Το Δεκέμβριο του 2012 προσδιορίσαμε δύο γραμμέ δράση. Πρώτον, έχουμε την αδειοδότηση για την Ευρώπη. Πρόκειται για διάλογο ανάμεσα σε όλου του εμπλεκόμενου φορεί που έχει ήδη ξεκινήσει, ούτω ώστε να καταλήξουμε συγκεκριμένε προτάσει και ένδικα μέσα για να αντιμετωπίσουμε τι ανησυχίε των καταναλωτών και κυρίω των νέων καταναλωτών. Ε, Φερρυπίν, δυνατότητα πρόσβαση πρόσβαση σε οπτικοακουστικό περιεχόμενο, όπως παραδείγματο χάρη το Catch Up TV, ε, σε διασυνοριακή βάση. Έχουμε κάνει πάρα πολλές συσκέψεις στην ομάδα εργασίας το τελευταίο εξάμεινο και σήμερα το απόγευμα εξάλλου θα έχουμε μια όλο μελή για την ενδιάμεση αναθεώρηση. Εκ παραλλήλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει την οικονομική και νομική αξιολόγηση του κεκτημένου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα του δημιουργού. Οι ενδεχόμενε πρωτοβουλίε που θα προκύψουν από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εδράζονται επί των αφισβήτη του εντοπισμού των προβλημάτων και των ενδεχόμενων νομοθετικών λύσεων που θα μπορούσαμε να δώσουμε σε Εργασίες που θα ξεκινήσουν με στόχο να λάβουμε απόφαση το 2014 για, για να καταθέσουμε προτάσεις νομοθετικού ε, μεταρρυθμιστικού σχεδίου. Δεν είναι ακόμη σίγουρο το τονίζω. Στη συνέχεια, η νέα αγορά τηλεπικοινωνιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με τη δική σας διάγνωση σχετικά με τις αδυναμίες της ενιαίας Ευρωπαϊκές Αγορές Τηλεπικοινωνιών. Ο η κυρία Βόρτμαν και ο κύριος Ρότ ξεκάθαρα το αναφέρουν αυτό στο ψήφισμά τους μετά από τις εργασίες που έκαναν. Έχει χάσει έδαφο ανταγωνισμός. Η Ευρώπη ε, στις τηλεπικοινωνίες ε, λόγω του παγκοσμίου ανταγωνισμού και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απίθυνε έκκληση για δημιουργία μια πραγματική ενίας αγοράς τηλεπικοινωνιών και θα συνεργαστούμε με στόχο να ε, εφαρμόσουμε ε, στην πράξη δύο βασικέ αρχέ συνθήκη λειτουργία Ευρωπαϊκή Ένωση, ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, τόσο ώστε όλοι οι πάροχοι να προσφέρουν ισότιμε υπηρεσίε σε όλου του καταναλωτέ, όπου και αν βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, ελευθερία για όλου του Ευρωπαίου και για τι επιχειρήσει να έχουν τι ψηφιακέ υπηρεσίε που επιλέγουν ανεξαρτήτω προελεύσεω. Ε, συγκεκριμένα, αυτά αποτελέσματα αυτό είναι ο στόχο μα. Ε, και ε, η Νέλη Κρός και σύσσωμη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές ε, του Σεπτεμβρίου και εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου αναμένεται να καταθέσει προτάσεις και θα είναι καταλητική σημασία η επικοδομητική υποστήριξη από πλευρά του Κοινοβουλίου. Ήδου, λοιπόν, Πρόεδρε, είναι προφανέ ότι η προτεραιότητα θα είναι ταχύστα να εγκρίνουμε τα ψηφίσματα που τώρα συζητούνται. Ε, θα μακροπρόθεσμα θα συνεχίσουμε το σχεδιασμό. Όλες τις προτεραιότητες τηλεπικοινωνιών θα τις προαγάγουμε και θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα θα οι συζητήσεις μας θα έχουν ιδιαίτερο βάρος για να μεριμνήσετε εσείς ούτως ώστε να υλοποιήσουμε τα υπεσχημένα από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, ε, τέλη Οκτωβρίου μάλλον αρχές Νοεμβρίου θα έχουμε εξελίξεις για την πράξη για την νέα αγορά ε, για να ενταθεί ε, ο δημόσιος διάλογος ε, για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου θα είναι εξαιρετική ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μπορέσει να εντοπίσει τους τελευταίους τομείς όπου χρειάζεται ανάληψη συγκεκριμένη δράση για να ολοκληρωθεί η ενιαία ψηφιακή αγορά πρώτου τέλους της παρούσης κοινοβουλευτικής θητείας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Τώρα θα περάσουμε στους ομιλητές που θα μιλήσουν εκ μέρους πολιτικών ομάδων. Η κυρία Σβάμπ δεν είναι μέσα στην αίθουσα. Ο κύριος Κορέια Δεκάμπος από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, θα ήθελα αρχίζοντας να ευχαριστήσω τον Επίτροπο διότι μας εξέθεσε όλες τις δυνατότητες που έχουμε για να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα προγράμματα, μας τα παρουσίασε εξάλλου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, τον Παύλο Άρες Εσκεβαρέ και τον Μάλκομ Χάρμπορ, όλος ιδιαίτερος, για το χώρο που δημιούργησαν, τόσο ώστε ε, με τη συνενετική εργασία να επιτύχουμε τους στόχους μας. Είναι καταπληκτικό το οικονομικό, δυναμικό αυτού του τομέα, το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει όσα του ότι ταυτόχρονα τονώνει την ανταγωνιστικότητα, την εγκύτητα των υπηρεσιών για τους καταναλωτές, ε, διότι υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες εναλλακτικές λύσεις ε, για τους καταναλωτές ε, και το ίδιο και για τους πολιτές και για τις επιχειρήσεις. Ηλεκτρονικό εμπόριο λοιπόν στα 28 κράτη-μέλη με 500 εκατομμύρια καταναλωτές. Τονώνεται έτσι το διασυνοριακό εμπόριο, καλύπτονται οι υπερπεριφερειακές ε, περιοχές ε, στο νησί του Κόρβου, στις Ασόρες, ε, μέσα στη μέση του Ατλαντικού, κοντά στις ΙΠΑ. Έχουμε το ρεκόρ των επιγραμμικών αγορών. Και στη συνέχεια βλέπουμε ότι με τις νέες ταχυδρομικές υπηρεσίες παραδίδονται βιβλία, έπιπλα, ε, ο κατάλογος είναι ατελείωτος. Με τις διασυνοριακές πωλήσει όμως πρέπει να κάνουμε και εμείς σημαντική πρόοδο. Ευρυζωνικές συνδέσεις, ε, ε, πρόσβαση σε ποιοτικά σύρματα δίκτυα, άρθρο 22 της οδηγίας για τους καταναλωτές όπου προβλέπεται μη διακριτική μεταχείριση ανάλογα με την χώρα στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση, κατοχυρώνονται ασφαλείς ηλεκτρονικές πληρωμές, τεχνολογική ουδετερότητα ως προς τις καινοτομίες και όλες τις σχετικές προκλήσεις, ε, δικαιώματα του δημιουργού, σήμα εμπιστοσύνη σε προϊόντα Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και γλωσσική φραγμή θα καταληθούν την ημέρα που θα καταφέρουμε να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη γιατί αυτό είναι λέξη κλειδί για τον 21ο αιώνα και την ε, ηλεκτρονική αγορά θα έχουμε κάνει ένα άλμα γίγαντα. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Φιώνα Χολ από το Άλντε. Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να χαιρετήσουμε την πρόοδο για την ε, ψηφιακή ενιαία αγορά, γιατί είναι ένα τομέα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει απτά αποτελέσματα στους πολίτες. Ε, στις αρχές εβδομάδας ε, είχαμε περαιτέρω μείωση του κόστους περιαγωγής. φοβερά νέα για φέτος, ε, τώρα που αρχίζουν και οι διακοπές. Αλλά όμως πρέπει να κάνουμε τα τελευταία βήματα και να δημιουργήσουμε μια πλήρως ανταγωνιστική ενιαία αγορά όπου οι τιμές ε, της περιαγωγής δεν θα υπάρχουν πια. Ε, θα πρέπει να υποστηρίξει η Κομισιόν την ε, ομάδα των φιλελεύθερων που είναι μπροστάρι σε αυτή την προσπάθεια. Θέλω να πω στου εκλογεί μου ότι θα σταματήσουμε να χρεώνουμε περιαγωγή. Όχι σε πέντε χρόνια, αλλά του χρόνου. Επίση, ελπίζω ότι μέχρι το επόμενο καλοκαίρι θα έχουμε κι άλλα καλά νέα για την ψηφιακή ατζέντα. Ελπίζω οι επιχειρήσει να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας ε, και στην ε, ε, σε ευρεία ζώνης υψηλής ταχύτητας. Ε, ούτως ώστε επίσης θέλω όλοι οι άνθρωποι με ειδικέ ανάγκες να μην αποκλείονται από τα ωφέλη της ψηφιακής εποχής και να είναι σε θέση να ε, δράξουν τα ωφέλη. Ελπίζω επίσης να, να μπορώ να καθησυχάσω τις επιχειρήσεις ότι η ευρωπαϊκή δράση αντιμετωπίζει το διασυνοριακό το κυβέρνιο έγκλημα. Ελπίζω, ελπίζω επίσης ότι οι μικρές επιχειρήσεις θα μπορέσουν να υποφεληθούν από αυτή την πρωτοβουλία. Όχι μόνο οι επιχειρήσεις ε, υψηλής τεχνολογίας, αλλά και οι υπόλοιπε. Θέλω και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις ε, ε επιτροπές οποιαδήποτε πόλη. Έχω ας πούμε ε, στην περιοχή μου ένα καφέ που κάνει δουλειές online και δίνει καφέ και διάφορα προϊόντα ας πούμε μέσω, που λιώνονται μέσω ίντερνετ. Χρειαζόμαστε τέτοιες δουλειές. Ελπίζω να, το... να μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα προς την ολοκλήρωση της ενίας αγοράς. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάλκομ Χάρμπορ από την ECR. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η ουσία της συζήτησης είναι ένα ψήφισμα για, από την Επιτροπή ε, Ενίας Αγοράς του Κυβουλίου. Εγώ, εγώ το πρότεινα ως πρόεδρος, όπου θέτει την ε, ψηφιακή ενία αγορά ε, στο κέντρο της προσπάθειας δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Και εγώ και ο Αντώνιο μίλησα, μίλησε για αυτό το θέμα. Πρόεδρε, να σας ρωτήσω γιατί μια και έχουμε ένα κοινοβουλευτικό ψήφισμα για αυτό το θέμα και οι συντάχτες οι συντάκτε δεν εκλήθησαν στην αρχή της συζήτηση. Ε, καλό θα ήταν λοιπόν ε, να έχουμε το σωστό πλαίσιο ας πούμε, και να εντάξουμε αυτή τη σημερινή συζήτηση στο πλαίσιο του ψηφίσματος. Η Επιτροπή ε, Ενίας Αγοράς ασχολείται με τις πολιτικές που χρειάζονται για να ε, ολοκληρώσουν την ενιαία ψηφιακή αγορά. εγώ και ο Παύλο Αρίας τους τελευταίους έξι μήνες ε, μαζί με άλλες ε, ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές έχουμε φτιάξει αυτά τα ψηφίσματα ο κ. Αρίας Δεκάμπος και τα Θέλω να ευχαριστήσω τις, τις άλλες επιτροπές πολιτισμού, απασχόλησης, νομικών υποθέσεων. υπέβαλαν σχόλια. Όπως είπε ο Επίτροπος, αυτό είναι πολύ περίπλοκο και επικύλο θέμα και χρειαζόμαστε ένα πολιτικό πλαίσιο για να προχωρήσουμε. Με τον ίδιο τρόπο που έχουμε ενθαρρύνει την ιδέα μέσω της ε, πράξης για την έννοια αγορά, έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Και χαίρομαι που είπατε ότι όταν γίνει η Σύνοδος Κορυφής θα προωθήσετε κάποιες δράσεις για την Σύνοδο αυτή του Οκτωβρίου. Ε, ε, το ψήφισμά μας έγινε ακριβώς για να σας ενθαρρύνουμε να το κάνετε πριν το καλοκαίρι. Το σημερινό μας μήνυμα και καλώ τους συναδέλφους να διαβάσουν ε, το λεπτομερές ε, ψήφισμα που ελπίζω να έχει την πλήρη υποστήριξη του, των Ευρωβουλευτών είναι ακριβώς αυτό. Καταληκτικά. Θέλω να πω αυτό που είπε η κυρία Χολ για τις ε, θέσεις απασχόλησης. Ήμουν την περασμένη εβδομάδα στην συνέλευση για την ψηφιακή ατζέντα, το ψηφιακό θεματολόγιο. Εκεί ακούσαμε πολλά παραδείγματα τέτοιου τύπου που μας είπε, όπως αυτό το καφέ, ας πούμε, στο Μπέρικ, όπου ε, ο κόσμος, ας πούμε, πλέον δουλεύει online, επιγραμμικά. Αυτό μπορεί να προωθήσει και την πρωτοβουλία για την νεολαία. Υπάρχουν ε, πολλά ελλείμματα στα ψηφιακά προσόντα μας. Ε, και έτσι θα τελειώσω, Πρόεδρε, με αυτό το σχόλιο. Αν χρησιμοποιήσουμε αυτά τα λεφτά για να βάλουμε τους νέους που έχουν αυτά τα προσόντα σε αυτές τις μικρές επιχειρήσεις, αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν να αλλάξουν μορφή, να μετασχηματιστούν, να αποκτήσουν νέα ορμή και η ευρωπαϊκή οικονομία δημιουργήσει περισσότερες, νέες, ε, περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Και σας παραπέμπω στη δουλειά που κάναμε στην Επιτροπή Ενίας Αγοράς. Ευχαριστώ κύριε Χάρμπορ. Ο κύριος Παύλο Αρία Ετσεβερία είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο κύριος Μάλκομ Χάρμπορ. Δεν ψηφίζουμε ακόμα ένα ψήφισμα στο Κοινοβούλιο. Ε, σε αυτή την νομοθετική θητεία κάνουμε πάρα ε, πολλές προσπάθειες για να υλοποιήσουμε αυτό το συγκεκριμένο στόχο. Και η επόμενη νομοθετική θητεία πρέπει, του Κοινοβουλίου θα πρέπει να ολοκληρώσει την ενιαία ψηφιακή αγορά, να ε, ολοκληρώσουμε αυτή την ε, ψηφιακή επανάσταση και να κάνουμε τα βήματα που χρειάζεται για να, την, να ολοκληρώσουμε αυτή την αγορά. Ο βασικός μας στόχος, όπως είπαμε και ε, στο κείμενό μας του Σεπτεμβρίου 2010, ήταν ακριβώς να ολοκληρώσουμε το ηλεκτρονικό εμπόδιο, η έκθεση του 12 Επίσης ε, λέει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε, ε, να ολοκληρώσουμε αυτή την αγορά. Δημιουργήσαμε και μια ε, ομάδα εργασίας που εδώ και δύο χρόνια έχει συνεδριάσει 26 φορές όπου συμμετείχαν 70 άτομα σε κάθε συνεδρίαση ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και του κλάδου και των βασικών οργανώσεων καταναλωτών και επιχειρήσεων. Πρέπει να τονίσουμε την παρουσία σε μία από αυτές τις συνεδριάσεις της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Επιτρόπου Μπαρνιέ στη συνεδρίαση του Ιουνίου του 2012. Αυτό το ψήφισμα βασίζεται στα, στις εργασίες που προέκυψαν από όλες αυτές τις συνεδριάσεις που σας ανέφερα και από την έκθεση επίσης που προανέφερα. Επίσης θα ψηφίσουμε κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ξεκινάμε μια δουλειά όπου ξεκίνησε με μια πρώτη κοινοβουλευτική δήλωση που μιλούσε για αυτή τη δέσμευση και που ζητούσε από τα άλλα θεσμικά όργανα, Κομισιόν και Συμβούλιο να κάνουν και αυτοί ό,τι πρέπει για να αναπτύξουν τι σωστέ πολιτικές, ούτω ώστε όλα αυτά να γίνουν πραγματικότητα. Ο επίτροπο μα έδειξε ότι έκανε πολλή δουλειά, ούτω ώστε όλα αυτά να γίνουν πραγματικότητα και ελπίζω ε, να δούμε και εμπράγματα τη δέσμευσή του. Νομίζω ότι μπαίνουμε στη τελική ευθεία, ούτω ώστε να φτάσουμε σε μια πραγματική ενιαία ψηφιακή αγορά. Σε όλη τη διάρκεια αυτή τη νομοθετική θητεία υιοθετήσαμε διάφορε προτάσει ε, νομοθετικέ για να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο. Και είμαστε σε φάση α, υλοποίησης όλων αυτών, τα δικαιώματα για τα, ε, την, ε, το cloud computing, προστασία ε, του δικαιώματος προσβασιμότητας, ε, τα δικαιώματα των καταναλωτών. Συνεχίζουμε τις προσπάθειες για να φτάσουμε σε μια πραγματική ψηφιακή αγορά στην Ευρώπη και θα συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες άοχνα. Γιατί πιστεύουμε ότι για να βγούμε από την κρίση πρέπει να προσπαθήσουμε ψηφιακά. Ευχαριστώ. Καλό όλους τους συναδέλφους να μην ξεπερνούν τον χρόνο τους παρακαλώ. Η κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. κινδυνεύουμε να εξαρτάται υπερβολικά πολλοί άνθρωποι από την ψηφιακή αγορά και να μείνουν ξεκρέμαστοι. Χρειαζόμαστε πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό χρειάζεται να είναι διασφαλισμένο. Χρειάζεται η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στο ίντερνετ υψηλή ταχύτητα, στην ουδετερότητα του διαδικτύου, στην ανάπτυξη ε, υποδομών. Αυτά είναι οι φράσεις κλειδί τις οποίες πρέπει να επεξεργαστούμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ρίας και τον κύριο Κορέα για την εξαιρετική τους ε, δουλειά σε αυτό το θέμα. Αυτά τα ερωτήματα είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντήσουμε. Η ουδετερότητα του διαδικτύου είναι μια βασική προϋπόθεση έτσι ώστε να μπορούν να διασφαλιστούν όλα αυτά τα πράγματα και γι' αυτό μου προκαλεί μεγάλη έκπληξη ότι το ΕΛΚ ακριβώς ε, για αυτό το σημείο ζήτησε χωριστή ψηφοφορία. Κύριε Σφάμπα, είδατε αυτό το αίτημα. Ευχαριστώ πολύ. Ορισμένε φορέ είστε και λογικό. Όπω έλεγα, η ουδετερότητα στο διαδίκτυο είναι κάτι θεμελιώδε, κάτι βασικό. Πρέπει να φροντίσουμε όλοι οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όλε οι επιχειρήσει, οι επιχειρηματίε να βρίσκονται σε αυτό το καθεστώς ίσης πρόσβασης. Ίση πρόσβαση λοιπόν με ίση ταχύτητα στο διαδίκτυο. Αυτό είναι σημαντικό, αυτό πρέπει να φροντίσουμε και πιστεύω ότι εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ καλό ψήφισμα και χαίρομαι για την ψηφοφορία που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σάκη, επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, η ενιαία αγορά είναι μια πολύ σημαντική κληρονομιά και ένας πολύ σημαντικός μύθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα όσον αφορά την ψηφιακή αγορά πρέπει να κινήσουμε γη και θάλασσα για να δώσουμε όθηση στην οικονομία. Οι προτεραιότητε του δημοσιονομικού πλαισίου αντιτίθεται σε αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ανταγωνιστική στην ψηφιακή αγορά. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο, χρειάζεται όμω πόρου για τον επόμενο αιώνα και όχι για τον αιώνα που τελείωσε. Ε, έχουν γίνει ουσιαστικές προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εναρμόνιση των ηλεκτρονικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Το υφισταμένο σύστημα είναι κατακαιρματισμένο, ιδιαίτερα όσον αφορά τον ε, γραπτό, τον έντυπο τύπο και πρέπει να επικαιροποιηθεί. Επίσης, η πρόσβαση στην πληροφορία πρέπει να είναι δεδομένη και να σταματήσει ο ανταγωνισμός στην ψηφιακή αγορά. Χρειαζόμαστε καινοτομία και ανταγωνισμό. Και πραγματικά ε, είναι ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να νομοθετήσει πλέον για την ουδετερότητα στο ίντερνετ, να προστατεύσει τους χρήστες. Οι πολίτες περιμένουν περισσότερα από τις κυβερνήσεις τους και δικαίως αυτό. Χρειάζονται πρότυπα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, για την ηλεκτρονική εκπαίδευση, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να αντιμετωπίζονται ίσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κίλαν, επόμενη ομιλήτρια. Η κινητοποίηση της ε, εσωτερικής αγοράς στον ψηφιακό τομέα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θα οδηγήσει, είμαι πεπισμένο, σε μια ανάπτυξη της ε, απασχόλησης. Χρειαζόμαστε ενισχύσεις όσον αφορά την ευρυζωνικότητα, την στήριξη των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στο ε, διαδίκτυο για τις διαδικτυακές τους δραστηριότητες. Χρειαζόμαστε ανταλλαγές στις εμπορικές πρακτικές. Πρέπει επίσης να προσέξουμε τις πολιτικές προτεραιότητες και να αποδομηθούν όλα τα εμπόδια. Τη διπλή φορολογία, οι διαφορές των ΦΠΑ για παράδειγμα και οι επενδύσεις είναι κάτι που χρειαζόμαστε ιδιαίτερα όσον αφορά την υποδομή σε πάρα πολλές περιφέρειες καθώς επίσης και καλύτερη οργάνωση των δικτύων και φυσικά διασφάλιση τη διαδικτυακή ουδετερότητα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε προγράμματα, χρειαζόμαστε βοηθητικά προγράμματα για να υποστηρίξουμε λοιπόν την ανάπτυξη τη ευρυζωνικότητα και στον, της των επιχειρήσεων στον τομέα του διαδικτυακού εμπορίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο Σβάμπ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, Πάμπλο Άρια και του κοιόδη εισηγητέ των, επόμενο, των υπόλοιπων ομάδων για αυτό το σχέδιο που έχουμε σήμερα στην Ολομέλεια. Η ψηφιακή εσωτερική αγορά, η ψηφιακή επανάσταση έχει πραγματικά δώσει όθηση στην ε, εσωτερική αγορά και οι καταναλωτές έχουν πλέον πολύ περισσότερες δυνατότητες. Αυτή η νέα πραγματικότητα που έχουμε, αυτές είναι δημιουργεί νέες προϋποθέσεις και νέες δυσκολίες είναι λοιπόν υποχρέωσή μα ιδιαίτερα στα πλαίσια τη ε, κρίση να δώσουμε βάση στην εξέλιξη της ε, ψηφιακή ενιαία αγορά για να την κάνουμε πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον λόγο αυτό, στόχο του ψηφίσματο μα είναι να προσπαθήσουμε μαζί να χαράξουμε το νέο πλαίσιο της ψηφιακής αγοράς έτσι ώστε όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να υποφεληθούν ε, από αυτό. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή επικρατεί κατακαιρματισμός νομοθετικός στην Ευρώπη η κυρία Τράουτμαν ξέρει ότι έχει εργαστεί σκληρά πάνω ακριβώς στο θέμα αυτό του κατακαιρματισμού και οι υπόλοιποι συνάδελφοι επίσης. Εγώ προσωπικά ε, ασχολήθηκα με την ε, οδηγία για την προστασία των καταναλωτών και πραγματικά όλες αυτές οι διαφορετικές νομοθεσίες που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα οδηγήσουν στο τέλος στην ε, παρεμπόδιση των καταναλωτών να κάνουν ηλεκτρονικό εμπόριο και πραγματικά πρέπει τα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν την νομοθεσία τους, να καταπολεμήσουν τα μονοπόλια και όσους επωφελούνται από αυτό ε, για το καλό των καταναλωτών. Επίσης, πρέπει να, καταστήσουμε σαφές πώς... το πώς μπορούμε να επωφεληθούμε από την ψηφιακή εσωτερική αγορά. Υπάρχει δυνατότητα αύξηση μέχρι 20% των εμπορικών συναλλαγών και μέχρι 15% όσον αφορά τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Ε, τα ηλεκτρονικά επίσης ε, καταστήματα θα οδηγήσουν σε μείωση του κόστους για τις ε, επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, κύριος Βάιντεν Χόλτσερ. Η ψηφιακή ενιαία αγορά είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση και την πρόθεση της ανταγωνιστικότητας. Έχει γίνει ε, φυσικά πρόοδος επάνω σε αυτό, όμως πραγματικά για να επιτευχθεί ο στόχος και να δώσουμε μεγαλύτερε μεγαλύτερες επιλογές και ευελιξία στους ε, καταναλωτές χρειάζεται προστασία της ε, ουδετερότητας, προστασία των προσωπικών δεδομένων και για μια, ομαλώς, για μια εσωτερική αγορά που λειτουργεί ομαλά χρειάζεται επίσης προσοχή στο περιεχόμενο. Χρειάζεται ίση πρόσβαση σε γρήγορες ευρυζωνικές υπηρεσίες για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Χρειάζεται επίσης η διασφάλιση ενός υψηλού επίπεδου συμμετοχής ε, από όλους στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Για να επιτύχουμε καινοτομία χρειάζεται η ανάπτυξη ενός ε, σαφούς και ξεκάθαρου συστήματος ε, πνευματικών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μακλάρκιν. Η ολοκλήρωση τη ε, ψηφιακή ενιαία αγορά πραγματικά θα ανοίξει πολλέ προοπτικέ στην ε, ενιαία αγορά και αυτό πρέπει να είναι μια κύρια προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ψηφιακή ενιαία αγορά θα μπορούσε να προσθέσει 800 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα. 420.000 δηλαδή ε, ευρώ περισσότερα για κάθε πολίτη. χρειάζονται ε, πολλές δράσεις. Ορισμένες από αυτές έχουν ήδη προταθεί για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, όπως, όπως για παράδειγμα τα κινητά δίκτυα ή κανόνες όσον αφορά τις ε, υπηρεσίες παράδοσης. Ωστόσο, με προβλημάτισε κάπω η πρόταση για το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των ε, πωλήσεων από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Δεν είμαι σίγουρη όσον αφορά ε, τα ωφέλη που θα έχει για τους καταναλωτές αυτή η πρόταση. Ωστόσο υποστηρίζω έντονα αυτό το ψήφισμα από του συναδέλφους μου και από τον συναδέλφο Μάλκομ Χάρμπορ. Είναι πραγματικά ένα πολύ καλό βήμα προ την ολοκλήρωση τη ενιαία αγορά. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντελκαστή Βέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω πιο, όσο πιο αποτελεσματικά μπορώ τα 90 δευτερόλεπτα που έχω. Θέλω να ευχαριστήσω τον Παύλο Αρίες, τον Μάλκομ Χάρμπορ για τις προσπάθειές τους. Οι πληροφόρεις, οι τεχνολογίες ενημέρωσης και επικοινωνίας είναι κινητήρη μοχλή για αυτή την προσπάθεια επί της οποίας εγκύπτουμε εδώ και 50 χρόνια και βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης, που είναι η ενιαία αγορά, η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Οι τεχνολογίες αυτές είναι ένας τρόπος για να διευκολύνουμε αυτή την προσπάθεια. Τα τελευταία πέντε χρόνια Αυτές οι τεχνολογίες ήταν κρίσιμες για να αναπτυχθεί περαιτέρω η ενιαία αγορά. Η ενιαία ψηφιακή αγορά είναι μόνο μία διάσταση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Θα ήθελα τώρα να εστιάσουμε σε κάτι που δεν νομίζω ότι το έχουμε αντιμετωπίσει και εξετάσει επαρκώς από εξετάσει επαρκώς όλοι όσοι δουλεύουν σε αυτόν τον τομέα πλήρης ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλη την Ευρώπη. Είναι κινητήριο μοχλός για ανάπτυξη. Αν εξασφαλίσουμε την πλήρη ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα, της δημόσιας διοίκησης σε όλη την Ευρώπη, τότε η ενιαία αγορά πραγματικά θα απογειωθεί. Κάμερε Βέρτ την επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Τρία πράγματα είναι σημαντικά για την ολοκλήρωση της ψηφιακής αγοράς από πλευρά σε πολιτισμού. Καταρχάς, το διαδίκτυο πρέπει να έχει ανοιχτό και δημόσιο χαρακτήρα. Χρειάζεται διασφάλιση της ψηφιακής, ε, της διαδικτυακής ε, ουδετερότητας ή διαφάνεια και οι προτάσεις που έχει κάνει η Επιτροπή δεν αρκούν. Δεν αρκούν σε καμία περίπτωση. Χρειάζεται επίσης να εγγυηθεί διαλειτουργικότητα και να προσέξουμε για την διαλειτουργικότητα. Αυτές είναι οι δύο βασικές ε, αρχές που πρέπει να διασφαλίζουν την ίση πρόσβαση σε όλους. Επίσης, πρέπει να είμαστε δημιουργικοί και να ενισχύσουμε την, τον τομέα των ε, πνευματικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο. Υπάρχει τεράστια πολιτισμική και οικονομική ε, δυνατότητα με την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Χρειαζόμαστε φυσικά πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για τα πνευματικά δικαιώματα στο διαδίκτυο και αυτό ευχόμαστε ως σοσιαλιστές. Επίσης, αποφασιστική σημασία για την ε, ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς είναι ότι ο καθένας πρέπει να έχει ίση πρόσβαση, να μπορεί εξίσου να χρησιμοποιήσει το ε, διαδίκτυο. Και εδώ πέρα χρειαζόμαστε υψηλά επίπεδα προστασίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πρόεδρε, Επίτροπε, η ανάπτυξη της ενίας ψηφιακής αγοράς είναι κρίσιμη για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών χωρών στις παγκόσμιες αγορές. Οι διαφορετικές τιμές, διαφορετικές υπηρεσίες, ίση άνηση κάλυψη, διαφορετικές ταχύτητες, ε, περίπλοκη σύνδεση ε, δημιουργούν προβλήματα στην λειτουργία της ε, ψηφιακής αγοράς. Θα χρειαστούν, θα υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση για μεταφορά δεδομένων και για το υπολογιστικό νέφος τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό θα πρέπει τα κράτη-μέλη να προσπαθήσουν να βρουν κοινέ λύσει σε αυτό το πρόβλημα. Πιστεύω ότι η ανάπτυξη ε, του ευρυζωνικού ε, διαδικτύου στα περισσότερα μέρη της Ευρώπης είναι προϋπόθεση για την πραγματική ενιαία ψηφιακή αγορά. Ε, προγράμματα υποστήριξης CEF α, της ευρείας ζώνης θα πρέπει να προωθηθούν. Εγώ ήμουν ε, και εισηγήτρια για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Χάντζλικ. Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντική η ενιαία ψηφιακή αγορά για την επιχειρηματικότητα. Έχουμε 27 διαφορετικά νομικά συστήματα και αυτό έχει υψηλό κόστος για τους επιχειρηματίες. Είναι πολύ δύσκολα αυτά τα εμπόδια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για τις επιχειρήσεις που δημιουργούν το 85% των νέων θέσεων απασχόλησης και αυτό συνέβη τα τελευταία πέντε χρόνια. Η ενιαία ψηφιακή αγορά είναι ευκαιρία για να μειωθεί η γραφειοκρατία, ε, για να διεθνοποιηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να βελτιωθεί το νομοθετικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν. Η Κομισιόν μίλησε επίσης για τη δυνατότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου και μίλησε για πρωτοβουλίες σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των πληρωμών, ας πούμε, στο ίντερνετ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις μικρομέσεις επιχειρήσεις που περιμένουν συγκεκριμένη δράση. Μία πλήρης ε, ψηφιακή αγορά θα δώσει ευκαιρίες για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχει τεράστιο δυναμικό που όχι μόνο θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε μια ισχυρή, ε, ζωντανή ε, οικονομία στο ίντερνετ, θα δώσουμε όμως και άλλες ευκαιρίες. Η ενιαία αγορά θα πρέπει καταρχάς να λειτουργεί σωστά, γιατί αλλιώς οι επιχειρήσεις δεν θα την εμπιστεύονται, δεν θα εμπιστεύονται τις ευκαιρίες ε, και δεν θα δραστηριοποιούνται οικονομικά εκεί μέσα. Επίσης πρέπει να δούμε την οδηγία για τις υπηρεσίες. Ε, η σωστή της εφαρμογή θα διευκολύνει την ανάπτυξη της ε, ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Συγχαρώ, ε, θέλω να συγχαρώ επίσης και τους εισηγητές. Ευχαριστώ κυρία Τχοτμάν. είναι η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όλοι θέλουμε να πετύχει η ενιαία ψηφιακή αγορά. Θέλω μόνο να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εργαλεία που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει με ε, πιο καλύτερο τρόπο ε, για τι τηλεπικοινωνίε. Θα μπορούσε να αρχίσει τονώνοντα ε, την αγορά, χρησιμοποιώντα τι αρμοδιότητες που έχει για την οριοθέτηση της διασυνοριακής αγοράς. Είναι ε, θεμελιώδη σημασία αυτό το εργαλείο, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σωστά. Κατόπιν, υποδομέ. Μας μιλήσατε για τις τηλεπικοινωνίες. Ο απολογισμός είναι θλιβερός. Ένα δις έχουμε για να εκπληρώσουμε στόχο ισότιμης πρόσβαση όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει ψηφιακή αγορά αν δεν έχουμε και τη δυνατότητα για όλες τις περιοχές, για όλους τους δήμους και κοινότητες, για όλους τους καταναλωτές να έχουμε ισότιμη πρόσβαση υπηρεσίες. Τρίτη και τελευταία παρατήρηση. Η συνολική θεώρηση δείχνει, ε, ε, ε, φαίνεται η βούληση του Κοινοβουλίου για να έχουμε μια συνεκτική πολιτική σε σχέση με τις επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της αγοράς καθώς και των καταναλωτών. Σας ευχαριστούμε. Μάζε Κούκοβιτς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τους συγητέ για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεση. Η ενιαία ψηφιακή αγορά θα διευκολύνει την ε, πρόσβαση και την λειτουργία των μικρομεσαίων υπηρεσιών, χαμηλώνοντας το κόστος λειτουργίας του. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό τα ο δημόσιος ε, τομέας να συμπεριληφθεί σε αυτήν την ε, μείωση του κόστους και αυτό θα οδηγήσει εν τέλει σε μείωση της φορολογίας για τους πολίτες. Η εσωτερική αγορά Επίσης θα μπορέσει να ε, προωθήσει τις ε, συνοριακές ε, διαδικτυακές υπηρεσίες υγείας και επίσης την εκπαίδευση και την διαβίου μάθηση. Επίσης και οι ηλικιωμένοι χρειάζονται και πρέπει να έχουν πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες. Δεν είναι μόνο οι νέοι οι οποίοι έχουν γεννηθεί με το διαδίκτυο αυτοί που το χρειάζονται. Χρειαζόμαστε λοιπόν ψηφιακά συστήματα, ψηφιακά μέσα τα οποία θα εγγυώνται την ασφάλεια των ε, δεδομένων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκάλο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όποιο και αν είναι ο τομέα δραστηριοτήτων, η χρήση της ε, ψηφιακής αγοράς είναι καταπληκτικό αναπτυξιακός πολλαπλασιαστής για τις επιχειρήσεις. Ακόμη για τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το να ενσωματωθούν τα νέα τεχνολογικά εργαλεία Του επιτρέπει να δρουν με αποτελεσματικότητα, ταχύτητα και εξοικονομώντα πόρου. Από αυτή την πλευρά πιστεύω θα έπρεπε να αναπτύξουμε μια πραγματική στρατηγική για το υπολογιστικό νέφος στην Ένωση, γιατί αυτό αντιστοιχεί στην τρίτη γενεά ε, της ψηφιακής τεχνολογίας ε, ε, ούτως ώστε να απελευθερωθούν οι υποδομές, ε, να μειωθεί το κόστος ε, χρησιμοποιώντας μηνιαία συνδρομή και μια διαρκή επικαιροποίηση των δικτύων. Πέρα από τις επιχειρήσεις, η ψηφιακή αγορά τροποποιεί και τις διαπροσωπικές σχέσεις των εργαζομένων σε σχέση με τους καταναλωτές. Οπότε δεν θα πρέπει να παραμελήσουμε τον ανθρώπινο παράγοντα. Οι Αμερικανοί φορείς ε, και με το Patriot Act ε, βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα χρησιμοποιώντας ε, συστήματα όπως το Prism για την παρακολούθηση και τις υποκλοπές. Αντίθετα, οι δικοί μας νομοί προστατεύουν την ακαιρεότητα και το απόρριτο των προσωπικών δεδομένων. Γι' αυτό αρμόζει να προκρίνουμε εγχώριους φορείς που διέπονται από τη δική μας νομοθεσία και άρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε να γίνουμε ανταγωνιστικοί να πτήσονται στις υπηρεσίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θα αρχίσει η διαδικασία Catch και έχουμε πέντε ομιλητές ε, ήδη. Η κυρία Ρουράτουν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε συζητήσει επί μακρόν το θέμα της ε, ψηφιακής αγοράς. Ε, έχουμε ακόμη πάρα πολλά να κάνουμε παρότι είχαμε μεγάλες επιτυχίες. Χαίρομαι που ο Επίτροπος Μπαρνιέ παρευρίσκεται στη συζήτηση. Τονίζω όμως ότι μόνο 6 από τα 10 ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν διασυνοριακές πωλήσεις. Είναι πολύ άριθμοι ακόμη οι φράγμοι. Συντελεστές ΦΠΑ παραδείγματος χάρη. Ε, ανεπαρκείς ταχυδρομικές υπηρεσίες. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμη να κάνουμε για να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, για να καταργήσουμε το κόστος περιαγωγής. Οι φιλελεύθεροι, τονίζω, δεν μας υποστήριξαν όταν θελήσαμε να μειώσουμε περαιτέρω το κόστος περιαγωγής. Αυτό που χρειάζεται κατά τη γνώμη μας είναι ε, αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους καταναλωτές και με τους επιχειρηματίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να χρησιμοποιήσουμε τον πλούτο της εμπειρίας του για να εξέλθουμε όλοι από την κρίση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θα ακούσουμε την κυρία Στάιλε. President, and thank you to Mr. Arias. Ευχαριστώ τον κύριο Αρίας και τον κύριο Ντεκάμπος για τη σημερινή συζήτηση. Συμφωνώ με την κυρία Γκέπχαρτ για την ε, ε, ψηφιακή ένταξη ε, με τον κύριο Κάστερ για το δημόσιο βίο. Γι' αυτό θα ήθελα να πω κάτι για τις ελευθερίες και την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά βιβλία, που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πολλές βιβλιοθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν πρόσβαση αυτή τη στιγμή σε βιβλία σε ψηφιακή μορφή, γιατί οι εκδότες αρνούνται να τους τα δώσουν σε ψηφιακή μορφή η γνώση δεν θα πρέπει να πληρώνεται. Στο κάτω-κάτω θέλουμε η οικονομία μας να βασίζεται υποτίθεται στη γνώση. Και αν θέλουμε να σταματήσουμε αυτό το apartheid των βιβλίων, χρειαζόμαστε συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή να αναλάβουμε δράση και πιστεύω ότι αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι βιβλιοθήκες θα έχουν βιβλία σε ψηφιακή μορφή, αυτό είναι απόλυτα εκ των Ουκάνευ για το, για το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Οι χρήστες του ίντερνετ, όπως επιβεβαίωσε και μία μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν χρησιμοποιούν όλη την ταχύτητα την οποία πληρώνουν στο διαδίκτυο χρησιμοποιούν μόνο το 1 τρίτον αυτή. Γι' αυτό λοιπόν η ευρυζωνία είναι κάτι σχετικό. Βέβαια, η ταχύτητα στο διαδίκτυο εξαρτάται από πολλά πράγματα, από τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, από τις δυνατότητες που έχουν τα καλώδια. Χρειάζεται όμως εγγύηση, αλλά εγγύηση για το εφικτό. Βέβαια, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σπάνια και συμβαίνει συνήθως στην Ήπεθρο οι συνδέσεις ε, διαδικτυακές να μην είναι γρήγορες και αυτό φυσικά επηρεάζει την ζωή και την ε, δραστηριότητα των ανθρώπων αυτών. Χρειάζεται λοιπόν καλύτερη υποδομή. Η μελέτη αυτή επίσης προτείνει ενίσχυση της ευρυζωνικότητας στην Ήπεθρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Γιασόφσκια. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Οι νέε τεχνολογίε παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση της ε, ψηφιακής οικονομίας. Ένα προσβάσιμο δίκτυο καθιστά δυνατό στους Ευρωπαίους να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί παγκόσμια. Το διαδίκτυο είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την αγορά, ιδιαίτερα όσον αφορά το διασυνοριακό εμπόριο και είναι ήδη σημαντικό από σήμερα. Χρειάζεται όμως επίσης να δούμε και τις ε, απειλές όσον αφορά τις ε, νέες τεχνολογίες επικοινωνίας ιδιαίτερα. Είναι πολύ σημαντικό να δραστηριοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταπολέμηση των ε, κινδύνων και να προωθήσει την δυναμική εξέλιξη της ευρυζωνίας στο διαδίκτυο. Επίσης χρειάζεται προσοχή όσον αφορά την διαδικτυακή απάτη, την εκλοπή ταυτότητας. Εκεί πρέπει οι κανόνες να αλλάξουν και να συνάδουν με τις εξελίξεις στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Σονκέλη. Συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, Όλοι οι συνομιλητές ετώνησαν την ανάγκη ολοκλήρωσης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Πραγματικά είναι κέρια σημασία για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι πολίτες έχουν ορθώς το δικαίωμα για ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα, για την πρόθεση του ηλεκτρονικού εμπορίου και για την ε, ίση πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα όπου και να βρίσκονται. Ιδιαίτερα όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι κάτι ζωτική σημασία. Χρειάζεται να ενθαρρύνουμε τους πολίτε να διεξάγουν περισσότερες εμπορικέ δραστηριότητε στο διαδίκτυο και τι επιχειρήσει να επίσης πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στην ασφάλεια τον Ιανουάριο άρχισε ένα πρόγραμμα το οποίο βοηθά τους νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις διαδικιακές τους δεξιότητες. Διότι αυτό μας λείπει και αυτό χρειαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σαρία, τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προσπάθειες που κατέβαλε και για το πρόγραμμα που υπέβαλε την περασμένη εβδομάδα. Η εσωτερική ψηφιακή αγορά για να εφαρμοστεί σωστά χρειάζεται να συμπεριλάβει τις ε, πληρωμές, τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Χρειάζεται να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ίση πρόσβαση σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης, ίση πρόσβαση με ίση ταχύτητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει ποιες αλλαγές θα διεξαχθούν στο, μέσο, στο μέλλον και πώς θα επηρεάσουν τις περιφέρειες στην Ευρώπη. Να πω επίσης ότι χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόταση αυτή. Ο κύριος Επίτροπος Μπαρνιέ δέχει το λόγο για να απαντήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω πολύ γρήγορα να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Σας άκουσα με μεγάλη προσοχή. Καταρχάς για να είμαστε σωστοί θα πρέπει να πούμε Πρόεδρε ότι συζητάμε σήμερα το πρωί την ε, εσωτερική ψυχιακή αγορά, γιατί το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς με τον Μάλκομ Χάρμπορ, με τον Αρία ε, Τσεβερία, έκανα μια τεράστια προσπάθεια με αυτό το ψήφισμα που είναι πολύ ακριβές, ε, ποικιλόμορφο, που υποστηρίζεται σχεδόν από όλους τους ευρωβουλευτές και από τις πολιτικές ομάδες και είναι μια ενθάρρυνση και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συνεχίσει τις προσπάθειές της. Θα ήθελα λοιπόν καταρχήν να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Χάρμπορ και τον Αρία Σετζοβερία. Με μεγάλη χαρά συμμετείχα στι εργασίε τη ομάδα πριν από λίγε εβδομάδε. Είναι ένα ψήφισμα αποφασιστική σημασία που διαφωτίζει τα βήματα που πρέπει να γίνουν ε, εφ' εξής. Και όπως είπατε κυρία Τρότμαν, ε, ίσως επιτέλους και χάρη στα πολλαπλά κείμενα τα οποία σας προανέφερα, αυτά που είχαμε, που φτιάχνουμε τώρα και που θα φτιάξουμε, ε, ελπίζω χάρη σε όλα αυτά λοιπόν να φτιάξουμε ένα σφαιρικό όλο για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Θα κάνουμε και άλλες ε, προτάσεις όπως σας είπα ε, στο επόμενο, στην επόμενη σύνοδο κορυφής του Οκτωβρίου. Πολλοί από εσά, ο κύριος Μπίελαν, ο πρώτος, ο κύριος Βάμπ, η κυρία Γκαλό, Μίλησαν για το υπολογιστικό νέφος. Ο κύριος Κέλλη μίλησε για τις επενδύσεις. Η κυρία Τότμαν ε, μίλησε για το Connecting Facility. Σας είπα και εγώ ότι δεν είναι επαρκής η πόρη που δίνουμε στο Connecting Facility. Νομίζω ότι σίγουρα πρέπει να επενδύσουμε στο ψηφιακό τομέα για να μην υπάρχουν διακρίσεις. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα των μη διακρίσεων. Γι' αυτό ακριβώς Ασχολήθηκα πολύ με την χρηματοπιστωτική ρύθμιση, με τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και πώς μέσω της νομοθεσίας και των ρυθμίσεων μπορούμε να ε, βοηθήσουμε ε, μέσω της διακυβέρνησης, μέσω της φορολογίας, μέσω πιστώσεων προφανώς, ε, μέσω της χρήσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων μπορούμε να προωθήσουμε τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις που χρειαζόμαστε για την ανάπτυξη αυτής της ενιαίας ψηφιακής αγοράς το Connecting Facility, το συνδέοντα στην Ευρώπη, το μέσο αυτό συνδέοντα στην Ευρώπη υπάρχει αλλά δεν αρκεί. Ε, κυρία Γκαλό μίλησε για το cloud. Ε, άλλοι μίλησατε για την προστασία των πολιτών ε, και τα προσωπικά τους δεδομένα. Και εγώ στην εισαγωγή μου είχα πει ότι αν υπάρχει ένα δίδαγμα μεταξύ άλλων που πρέπει να βγάλουμε από αυτή την κρίση για την ε, κατασκοπία των Αμερικανών επί της Ευρώπης, είναι ότι στο μέλλον πρέπει να δείξουμε μια πολιτική βούληση, ούτω ώστε η Ευρώπη να έχει εργαλεία για τη στρατηγική αυτονομία της. Γαλιλαίο, ε, τηλεπικοινωνίες, αλλά και το υπολογιστικό νέφος, σαφώς, το cloud computing. Και αυτό είναι τμήμα αυτής της στρατηγικής. Έχουμε διάφορα εργαλεία σε όλους αυτούς τους τομείς για να φτιάξουμε αυτή την, την στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Να τη χτίσουμε, να την οικοδομήσουμε. Κυρία Τροτμάν, μίλησε για την δράση που προωθούμε για να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα την νομοθεσία που υπάρχει της τηλεπικοινωνίας. Οι δράσεις μας βασίζονται στο, στην πραγματικότητα, την ανταγωνιστική των αγορών, που δυστυχώς ακόμα είναι πολύ εθνική, πολύ κατακαιρματισμένη. Ε, η πρωτοβουλία που παρουσίασε η κυρία Κρούζ το Σεπτέμβριο για τις τηλεπικοινωνίες ακριβώς καλύπτει αυτά τα κενά με την υποστήριξή σας, ούτως ώστε να φτιάξουμε μια πραγματική ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Πολλοί από εσά μίλησαν για το θέμα των διακρίσεων και την ανάγκη πρόθεση των μη διακρίσεων. Κυρία Κορέα Ντεκάμπο, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν αυτές οι περιφερειακές υπερπόντιες περιοχές, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Ε, υπάρχουν διακρίσεις λόγω απομάκρυνσης, απομόνωσης κάποιων περιοχών. κυρία Γκέπχαρτ, η κυρία Μαϊζέκοβιτς μίλησαν και, και αυτές για αυτό το θέμα. Δεν ξεχνώ επίσης αυτό που υπόθηκε για την διάκριση λόγω ηλικίας, διαφοράς γενιάς. Σωστά επιμένετε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν γεωγραφικές διακρίσεις ε, των καταναλωτών. Γι' αυτό θα δημοσιεύσουμε έναν οδηγό για την εφαρμογή αυτής της αρχής με βάση το άρθρο 20 της Οδηγίας ε, για τις Υπηρεσίες. Κυρία κυρία, κύριε Βάιντεν Χόλτσερ, κυρία Κάμερβερ που μίλησατε για τα δικαιώματα των δημιουργών. Η δουλειά που κάνω εδώ και τρία χρόνια προωθεί διάφορα κείμενα στο Συμβούλιο που δεν έχουν ακόμα ψηφιστεί. Ο σκοπός είναι τα δικαιώματα των δημιουργών να εξυγχρονιστούν, να, εξυγχρονιστούν, να ενταχθούν στην εποχή μας ίντερνετ, ε, ούτως ώστε οι περισσότεροι ε, καταναλωτές να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο που θέλουν. Επίσης για τις άδειες τις πολυεδαφικές που θα, θα τις έχουμε προσεχώς, ούτως ώστε να έχουμε καλύτερη διαχείριση των δικαιωμάτων των δημιουργών. Η Φιώνα Χολ, η Ροζατούν μίλησαν για το θέμα της περιεγωγής. Την 1η Ιουλίου είχαμε μια νέα μείωση των τιμών της περιαγωγής. Θα πρέπει προφανώς να πάμε ακόμα πιο μακριά. Αυτή η πρωτοβουλία που ετοιμάζουμε τις λεπικοινωνίες που μόλις ανέφερα, ε, όπως είπε και η Νέλη Κρούς, ε, τελικά η υπερχρέωση της περιαγωγής θα ε, εξαφανιστεί. Ε, μας είπατε κυρία Χόλ ότι πρέπει να επισκεφτούμε και αυτό το ψηφιακό καφέ στην ε, δική σα εκλογική περιφέρεια. Όταν έχω χρόνο να βγω από το γραφείο μου, με μεγάλη χαρά θα έρθω σε εσά να σε επισκεφτώ. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Κυρία Γκέπχαρτ. Κύριο Σάρκε. Κυρία Σάκε. Μίλησε για τις υποδομές ε, τις η ουδετερότητα του δικτύου είναι πολύ σημαντική, καθώς και η καθολική πρόσβαση στις ευρυζωνικές, στο ευρυζωνικό διαδίκτυο. Το Connecting Facility θα συνεισφέρει σε αυτό και ε, επίσης αυτή η πρωτοβουλία για την ουδετερότητα του δικτύου προωθείται φέτο, υπό την αιγίδα της Νέλης Κρούς. Ε, νομίζω ότι θα βοηθήσει σε αυτό. Για τα ανοιχτά πρότυπα που ανέφερε η κυρία Σάκε. Και εδώ θα διευκρινίσουμε τη θέση μας και πρέπει να προωθήσουμε αυτό που επιθυμείτε κι εσείς, ανοιχτή πρόσβαση μέσω αυτών των προτύπων. Η Κομισιόν μόλις υιοθέτησε μία ανακοίνωση για αυτά τα πρότυπα, κυρίως στο πακέτο τηλεπικοινωνιών. Η κυρία Κάθλιν μίλησε για τα κοινά δικαιώματα πώληση και εξέφρασε αμφιβολίες. Ε, θα είναι προαιρετικό κάτι τέτοιο. Ο, ο έμπορος μπορεί να πουλάει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με υψηλό επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές δεν αντικαθιστούμε τους εθνικούς κανόνες και νόμους για την κατανάλωση, απλώς είναι μια επιπλέον επιλογή που έχουμε, που δίνουμε μάλλον. κυρία Χάντσλικ, κυρία Δεκαστή Βέρα, μίλησαν για κάτι πολύ σημαντικό, ε, επί των οποίων μπορούμε να κάνουμε εξοικονόμηση χάρη στην ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, του δημόσιου τομέα. Είναι το 18% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ αυτό. Και θέλω να πω για αυτό το θέμα ότι έχω παρουσιάσει πολλέ πρωτοβουλίε με του συναδέλφου μου ακριβώ για να προωθήσουμε αυτή την ψηφιοποίηση. Πρόσφατα η ηλεκτρονική υπογραφή, ακόμα πιο πρόσφατα η ηλεκτρονική τιμολόγηση. Θα ήθελα μαζί με σας να καταφέρουμε αυτή την ε, ψηφιοποίηση. Υπάρχουν 90 ε, δισεκατομμύρια ε, ευρώ που μπορούμε να εξοικονομήσουμε κάθε χρόνο αν ξεφορτωθούμε τη χαρτούρα χάρη στην ψηφιοποίηση. Τελειώνοντας, κυρία Στήλερ, ε, μιλήσατε για το πρόβλημα, την πρόκληση των ψηφιακών βιβλίων. Η Κομισιόν ήδη έχει αναλάβει δράση σε αυτό το θέμα, ούτω ώστε να εμποδίσει τι περιοριστικέ πρακτικέ. Ο κ. Σαλμούνια το προωθεί αυτό. Αυτή η αγορά αναπτύσσεται και υποστηρίζουμε αυτό το κίνημα με πολλέ στρατηγικέ αυτό περιμένω από την ε, πρωτοβουλία Licensing Europe, αδειοδοτώντας την Ευρώπη. Σήμερα το απόγευμα θα κάνουμε την ενδιάμεση αξιολόγηση αυτής της προσπάθειας και πραγματικά περιμένω να δω τα αποτελέσματα των διαφόρων ε, ε, εργαστηρίων που έχουμε ανοίξει για αυτό το θέμα για να δούμε τι πρόοδο έχουμε σημειώσει. Η πρωτοβουλία μας, όπως είπε ο κ. Σαρίας, πρόσφατα, ε, σύντομα θα έχει και πρωτοβουλίες για τη διακυβέρνηση. Και θα προσέξω πολύ τις προθεσμίες που χρειάζονται, ούτως ώστε να υλοποιήσουμε τους στόχους που θέσαμε για όλα αυτά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κυρίως τους δύο προτεργάτες αυτού του θέματος, τον Μάλκομ Χάρμπορ και τον κύριο Αρίας Τσεβερία, για τη δέσμευσή τους, πολύ χρήσιμη για μας. Όλα αυτά τα έχουμε συγκεντρώσει το, στο ψήφισμά σα βλέπουμε ότι τα θέματα και οι άξονε είναι πολύ άριθμοι, αλλά νομίζω ότι έχουμε μια σφαιρική εικόνα για αυτό το τεράστιο εργοτάξιο που είναι η νέα ψηφιακή αγορά. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Έχω το επόμενο σχέδιο ψηφίσματος. 73-331 του 2013 από την Επιτροπή